Ευχαριστούμε πολύ. Πριν ε, να τελειώσουμε, έχω μια ανακοίνωση. Από την ομάδα των φιλελεύθερων μου έχει ζητηθεί να ορίσω τον Γιβένε Μαρίνη όσον να αντικαταστήσει τον ε, Τζαμάρο Ούγκιας που ήταν στην Επιτροπή Μεταφορών και αντικαθιστά τον Βιτσέντσο Ιωβίνε. Υποθέτω ότι εγκρίνεται, αφού δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Συνεπώς,